Κυρίε Κυρίες και κύριοι, καθίστε, δεν χρειαζόμαστε απαρτία. Είναι ελάχιστη παριστάμενη το ακροατήριο, αλλά βλέπετε έχουμε εκπομπή στο διαδίκτυο. Και έτσι αποφασίσαμε να συνεχίσουμε με τα σημεία της ημερήσιας διάταξης. Καλωσορίζω λοιπόν τον κύριο Γκαμπόρ Ιγκλώτη, διευθυντής αρμόδιος για τη διαχείριση των κρίσεων. Δηλαδή είναι ένας φορές ανάμεσα σύνδεσμος μετα... εντός του... της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσεως. Θέμα μας είναι η διαχείριση των κρίσεων από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλωσορίζω τον κύριο Ικλόντι θα τον παρακαλέσω να προβεί σε κάποια προκατακτικά σχόλια και είμαι σίγουρη ότι θα είναι ενδιαφέροντα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για την εισαγωγή σας. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και που περνάω το απόγευμά μου μαζί σας. Για μία ώρα, ίσως λίγο παραπάνω. Ήδη έγινε ανταλλαγή απόψεων σήμερα με τον Water Stevens που είναι πρόεδρος της Επιτροπής για την Πολιτική και την Άμυνα και κάλεψε ευρύ φάσμα θεμάτων θέματα που απασχολούν την Επιτροπή αυτή, αποστολές, επιχειρήσεις. Πριν έρθω εδώ είχα τη δυνατότητα να ρίξω μια ματιά στις σημειώσεις του ούτως ώστε να είμαι σίγουρος ότι δεν θα επαναλάβω αυτά που σας είπε ήδη. Και ακόμα χειρότερα μην πω τίποτα που είναι εντελώς αντίθετο με αυτά που είπε. Με βάση αυτό θα έλεγα ότι έχετε μια καλή εικόνα για το που βρισκόμαστε όσον αφορά τις αποστολές, τις επιχειρήσεις και τα βασικά ζητήματα που μας απασχολούν και η πρόσφατη ακρόαση του νέου υπατου εκπροσώπου της κυρίας Μογκερίνης νέας υπάτου εκπροσώπου την περασμένη εβδομάδα τον περασμένο μήνα συγγνώμη Ακούσατε επίσης και μια αποτίμηση της ΚΕΠΑ, ποιες ήταν οι επιτυχίες, ποιες ήταν οι αποτυχίες και πώς θα ήθελα να προχωρήσουμε από εδώ και εμπρός. Δεν θα προσπαθήσω να επαναλάβω τα μηνύματα που σας έδωσε. Είναι η πρώτη δυνατότητα που έχω να έρθω εδώ και να συναντηθώ μαζί σας, αλλά έχω ελπίδες ότι πολλές ε, συναντήσεις θα ακολουθήσουν. Να πω ευθύ εξ αρχής ότι εγώ και η διεύθυνσή μου, η αρμόδια για την ΚΕΠΑ είναι, αρχική, είναι ανοιχτή υπεύθυνη για την ΚΕΠΑ μάλλον, να σας βοηθήσει στις καθημερινές σας εργασίες. Είμαστε προσβάσιμοι, ανοιχτοί με τα χαράς να επανέλθω και άλλη μια φορά, να έρχομαι τακτικά αν θέλετε, όποτε είναι αναγκαίο και αν υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα που προκύπτουν στις συζητήσεις με τα χαράς να σας δώσουμε τις αναγκαίες πληροφορίες και να συζητήσουμε και πληροφορίες που χρειάζεται και εσείς για να συζητήσετε μεταξύ σας. Σας χρειαζόμαστε. Πρέπει να είσαστε πάντα ενήμεροι. Να ξέρετε τι έχει δρομολογηθεί και τι πρόκειται να δρομολογηθεί. Θέλουμε να σας ενημερώνουμε. Να σας ενημερώνουμε και για αυτά τα θέματα που βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού. Θέλουμε να ξέρουμε και τις δικές σας απόψεις για διάφορα ζητήματα. Και τέλος, εξίσου σημαντικό, χρειαζόμαστε τη στήριξή σας. Άρα είναι αμφίδρομος η διαδρομή με τα χαράς να σας βοηθήσουμε στις καθημερινές εργασίες σας, αλλά χρειαζόμαστε και την υποστήριξή σας και την κατανόησή σας. Όπως είπε και η κυρία Πρόεδρος, εργαζόμουν λοιπόν από τον Ιούνιο στην υπηρεσία για πέντε μήνες στη μονάδα για διαμόρφωση της πολιτικής και έπρεπε και εγώ να προσπαθήσω να προλάβω τις γρήγορες αλλαγές του περιβάλλοντός μας. Να πω λίγα λόγια για το πρόσωπό μου. Ήμουν διπλωμάτης ε, πάνω από 30 χρόνια στην Ουγγρική Υπηρεσία Εξωτερικών, τελευταία μου θέση, ήταν στο ΝΑΤΟ. Ήμουνα βοηθός γενικός γραμματέα για θέματα τα οποία είναι νέα για το ΝΑΤΟ. Αναδιόμενες προκλήσεις για την ασφάλεια ο τίτλος. Κυβέρνοτρομοκρατία, πυρηνικά θέματα, θέματα διάδοσης πυρηνικών όπλων κλπ. Και αυτά θα με βοηθήσουν και στην παρούσα μου ιδιότητα. Uh, uh, to tell you a few Κάτι για τη μονάδα μου, την ίδια ίσως να μην γνωρίζετε ακριβώς την υπηρεσία μου και ποια εντολή έχει αναλάβει. Να πω μερικά λόγια για τις μεγάλες προτεραιότητές μας. Uh, then, κρίσεων, αποστολές, επιχειρήσεις, Μερικά λόγια για τις ε, εταιρικές σχέσεις που γίνεται όλο και πιο σημαντικό στοιχείο στην καθημερινή μας δουλειά, συνεργασία και με άλλους διεθνείς οργανισμούς αλλά και με χώρες εταίρους και κάποια διλήμματα. Να σας δείξω κάποια διλήμματα uh, που βρισκόμαστε με τις αποστολές και τις επιχειρήσεις όπου εκεί δεν υπάρχει μια σαφής ε, θέση ναι, θα ήθελα να γνωρίζετε να καταλάβετε ποια είναι τα διλήμματα και όλα αυτά για να μπορέσω να σας δώσω μια καλύτερη εικόνα. Ξεκινώντας με, την, με το CSPD είναι αφορά τον σχεδιασμό, την αντιμετώπιση των κρίσεων και το σχεδιασμό. Crisis Management and Planning. Είναι μια υπηρεσία εντός της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης και είναι στο επίκεντρο της κοινή ασφαλείας και της άμυνας και της σχετικής πολιτικής δημιουργήθηκε δημιουργήθηκε το 2009 μετά συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κορυφής που ήθελε να δημιουργηθεί μία νέα ένα στρατηγικό σχεδιασμό συμπεριλαμβάνει και τον πολιτικό τομέα και το στρατιωτικό για επιχειρήσει τη κοινή πολιτική άμυνα και ασφαλεία. Μιλάμε για στρατιωτικέ επιχειρήσει και μιλάμε για αποστολέ που είναι πολιτική φύσεω αποστολέ. Βλέποντας λοιπόν την εντολή του CMPD ε, θέλουμε να κάνουμε στατηγικό αρχικό σχεδιασμό των αποστολών και των επιχειρήσεων. Θέλουμε την επόμενη περίοδο να τονίσουμε περισσότερο το τελευταίο κομμάτι, δηλαδή την εκ των προτέρων, τον εκ των προτέρων σχεδιασμό, ώστε να μην υποχρεωθούμε να ασχοληθούμε με τις συνέπειες της κρίσης, αλλά να μπορούμε εκ των προτέρων να σχεδιάζουμε και να μπορούμε να δίνουμε επιλογές εκείνους που παίρνουν τις αποφάσεις. Ε, να ξέρουμε ποιες είναι οι ενδεχόμενες δράσεις που μπορούμε να εφαρμόσουμε, τι πόρους έχουμε και ποιες είναι οι διάφορες συνέπειες των διαφόρων αποφάσεων. Επίσης έχουμε το ρόλο του συντονισμού, της δημιουργίας δυνατοτήτων και στην πολιτική πλευρά και στην ε, στατιωτική. Όπως γνωρίζετε από τη στατιωτική πλευρά ο βασικός που κινείται και δρά είναι η EDA, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Αμήνη. Ασχολείται κυρίω με την ανάπτυξη δυνατοτήτων στο δυτικό τομέα. Εμεί θα πρέπει να μπορούμε να εναρμονίζουμε τι προσπάθειε και να συντονίζουμε. Συντονίζουμε τι προσπάθειε μεταξύ πολιτικού και στρατιωτικού τομέα. Έχουμε ευθύνε στον τομέα τη ΚΕΠΑ για συμπράξει όπως ανέφερα, αυτό είναι κάτι που αυξάνεται συνεχώς. Έχει όλο και μεγαλύτερη σημασία. Και προβαίνουμε και σε σεμινάρια, καταρτήσεις. Έχουμε το Κολέγιο για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα που ανήκει στην Διεύθυνση Διαχείρισης Κρίσεων και Σχεδιασμού και συνεργαζόμαστε να πετύχουμε καλύτερους στόχους και θέλουμε να αναπτύξουμε ε, διάφορες έννοιες και σχέδια ξεκινώντας το διάστημα, ε, να βρούμε τι γίνεται συνεργασία μεταξύ ασφαλείας και θεμάτων εσωτερικών και δικαιοσύνης. Να πω κάτι για τις βασικές προτεραιότητες που βρίσκονται μπροστά μας. Θα ξεκινήσω αναφερόμενος το Συμβούλιο του 2013, του Δεκεμβρίου του 2013, τη Συνόδο Κορυφής, που θα θυμόσαστε, έθεσε, εκεί τέθηκε καν οι βάσεις για τη συζήτηση ε, θεμάτων αμήνης. Ήταν ε, πάρα πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή και λάβαμε έναν κατάλογο καθηκόντων για μια επόμενη πενταετία από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Συμπεριλαμβάνονται 60 συνιστώσεις. Δεν είναι όλα τα σημεία και τα καθήκοντα εκείνα για τα οποία εμείς ηγούμεθα, αλλά σε αρκετούς τομείς, στους περισσότερους, εμείς πρέπει να ηγηθούμε των προσπαθειών. Πρέπει να δίνουμε λόγο, να δώσουμε λόγο στο, στη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου, δηλαδή 1,5 χρόνο μετά την ανάθεση των καθηκόντων. Όταν λέω ότι από τα 60 καθήκοντα είχε τεθεί σαν όριο χρονικό Ιούνιος 2015 δεν σημαίνει ότι πρέπει να περιμένουμε μέχρι τον Ιούνιο του 2015 για να κάνουν πράγματα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση πριν τον Ιούνιο του 2015 ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε το φάσμα θεμάτων όπου χρειάζεται να το συζητήσουν οι κρατών και κυβερνήσεων. Να συζητήσουν τρία-τέσσερα θέματα οι των και κυβερνήσεων. Αν παραμείνουν μπροστά τους περισσότερα ζητήματα, θα είναι σχεδόν ανέφικτο να περιμένουμε από αυτούς να λάβουν σημαντικές αποφάσεις και να προχωρήσουν. Ήδη αυτό το Νοέμβριο στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Αμήνης θα υπάρξει δυνατότητα να ξεκινήσει η εξέταση των θεμάτων και να βγάζουμε από τη μέση κάποια ζητήματα. Έχουμε, ε, έχουμε ξεκινήσει ήδη κάποιες προσπάθειες, παραδείγματος χάρη για πρώτη φορά θεσπίζεται μια, θεσπίστηκε τον Ιούνιο μια στρατηγική ε, για τις Ευρωπαϊκές Ενώσεις για, τα, για τη θάλασσα, το θαλάσσιο τομέα. Και θα μας δώσει και σχέδιο δράση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή τελικά πώς θα εφαρμοστούν τα λόγια, πώς θα υλοποιηθούν τα λόγια της στρατηγικής στην πράξη. Το Συμβούλιο Εξωτερικών και Αμήνης του Νοεμβρίου φέτος θα υθετήσει ελπίζω ελπίζω, συμπεράσματα για θέματα όπως η πολιτική αμήνη στον κυβερνοχώρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και πιο σχετικό πλαίσιο ή για αμυντική συνεργασία ή χρηματοδότηση στατιωτικών αποστολών που δεν είναι και κάτι εύκολο, είναι επίμαχο ζήτημα. Και τώρα και στο προβλέψιμο μέλλον πιστεύω ότι έτσι θα είναι. Υπάρχουν κάποιες νέες πρωτοβουλίες οι οποίες ανετέθησαν από το Συμβούλιο Κορυφής του Δεκεμβρίου. Τελικά αποτελέσματα δεν θα παρουσιαστούν στη συνεδρίαση του Νοεμβρίου ε, αλλά μπορούμε να κάνουμε μια αποτίμηση, να πάρουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές και να συνεχίσουμε. Να αναφέρω ένα θέμα από τα βασικά στοιχεία εκπαίδευση και εξοπλισμός. Είναι πιλωτικό πρόγραμμα και να αυξηθούν οι δυνατότητες. Enable and enhance. Να δώσεις περισσότερες να δώσεις δυνατότητες και να διευρυνθεί το πεδίο των δυνατοτήτων σε ελεύθερη μετάφραση. Στόχος είναι σαφής να δώσουμε δυνατότητα σε χώρες και περιφέρειες που είναι μακριά από την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να έχουν τη δυνατότητα οι ίδιες να αντιμετωπίσουν προβλήματα που παρουσιάζονται στη γειτονιά τους ή στην επικράτειά τους. Αντί να πρέπει να περιμένουμε πρόσκληση να παρέμβουμε και να στείλουμε αποστολές και να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της κρίσης. Αναφερόμαστε σε τρία θέματα. Και η εμπειρία μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να τεθεί προτεραιότητα σε αυτά τα θέματα. Η δυνατότητα, η δημιουργία δυναμικού θα γίνεται κάτι όλο και πιο σημαντικό στο έργο για τη διαχείριση των κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι μόνο στην περίπτωση που ήδη υπάρχει κρίση, αλλά θέλουμε να έχουμε προσέγγιση αποφυγής των συγκρούσεων να επιτρέπουμε σε περιφερειακές, ε, περιφερειακούς οργανισμούς όπως η Αφρικανική Ένωση να κινηθούν, να έχουν την κατάρτιση, να μπορούν να κάνουν την ε, δουλειά τους επιτόπου. Εκεί που μπορεί να κινηθεί η Φερρυπίνη η Αφρικανική Ένωση. Ήθελα να προσθέσω κάτι το οποίο είναι εμπειρία πρακτική. Από μόνη της η εκπαίδευση δεν αρκεί. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Όπως ε, της αποστολής στη Λιβύη. Εάν δεν δώσουμε τον αναγκαίο εξοπλισμό σε εκείνους που έχουν εκπαιδευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και ίσως μπορεί να, να και άλλα ας πούμε μηχανήματα για την τηλεπικοινωνία για, χρειάζονται τα κιάλια για τον έλεγχο των συνόρων στη Λιβύη, Φερρυπίν. Ε, για να τα λέω ξεκάθαρα τα πράγματα μεταξύ μας, πρέπει να προσπαθήσουμε τους ντόπιου να τους προσελκύσουμε στη διαδικασία. Αν δώσουμε τον αναγκαίο εξοπλισμό θα ενδιαφέρονται περισσότερο. Αν πάμε εκεί και τους εκπαιδεύουμε απλώς και δεν τους δίνουμε τίποτα, ανάλογα με τη χώρα και τις περιστάσεις ε, εξαρτάται και η αντίδραση και οι στόχοι δεν θα επιτυγχάνονται. Ο εξοπλισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και τι το στοιχείο, βιωσιμότητα, ε, πολύ σημαντική. Να αναφέρω ένα παράδειγμα από το ΝΑΤΟ, το ISEF. 350.000 στρατιώτες εκπαιδευτήκαν, αφήσαμε εξοπλισμό πίσω μας για να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά εάν δεν μέναμε να είμαστε σίγουροι ότι ο εξοπλισμός μπορεί να συντηρηθεί, τότε το φορτηγό θα λειτουργούσε όσο είχε καύσιμα, ο εξοπλισμός θα χρησιμοποιείται μέχρι να σπάσει κάτι και λήψη ανταλλακτικών, ο εξοπλισμός θα είναι άχρηστος και θα είναι πεταμένα χρήματα και θα χρησιμοποιείται. Βιωσιμότητα είναι πάρα πολύ σημαντική στη διαδικασία και θα επανέλθω σε αυτό το ζήτημα για να στείλω ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Όλες αυτές οι προσπάθειες είναι μακροπρόθεσμες από τη φύση τους. Καμία δεν είναι βραχυπρόθεσμη. Είναι λανθασμένη η αντίληψη ότι αυτές οι προσπάθειες είναι βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα. Αλλάζει η μορφή ενδεχομένως, αλλά η προσπάθεια θα πρέπει να διατηρείται, να είναι βιώσιμη. Αυτά λοιπόν για την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό. Έχουμε κάποια κρίσιμα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα έχουμε το πρόβλημα, την πρόκληση για τον εξοπλισμό. Και το άλλο είναι η χρηματοδότηση. Η πρόκληση όσον αφορά τον εξοπλισμό, το πρόβλημα του εξοπλισμού σε μεγάλο ποσοστό αφορά το είδος του εξοπλισμού. Μιλάμε για μη θανατηφόρο ε, εξοπλισμό διπλής χρήσεως ή και φωνικά όπλα και φωνικό εξοπλισμό βλέπουμε πώς θα εξελιχθούν οι συζητήσεις. Αλλά εν γέννη θα συγκεντρωθούμε σε μη φωνικό εξοπλισμό και ίσως κάποια στοιχεία εξοπλισμού διπλής χρήσεως και τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στα διαφορα κάτι κράτη-μέλη. Όπως Ιράκ και βοήθεια προς τους Κούρδους, να ένα παράδειγμα. Δεν είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να δώσει πυρομαχικά εξοπλισμό στους Κούρδους. Τα κράτη-μέλη μπορούν να το κάνουν και το κάνουν και το κάνουν αυτό. Αλλά προσπαθούμε να επεκτείνουμε τα όρια μας όσον αφορά την χρήση των χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να δίνουμε τις ικανότητες που απαιτούν αυτές οι χώρες για να α, μην επιδεινώνεται η κρίση. Να αποφεύγουμε επιδεινώσεις. Προβλέπω τρία διαφορετικά ενδεχόμενα. Συγγνώμη που μιλάω τόσο πολύ γι' αυτό, αλλά είναι βασική έννοια αυτή, βασική. Λοιπόν, υπάρχει μια κρίση, ας πούμε. Εκτελούμε μια αποστολή για διαχείριση της κρίσης. Εκπαιδεύουμε τις δυνάμεις, εξοπλίζουμε τις δυνάμεις, ούτως ώστε να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να φύγουμε εμείς. Όπως στο Μαλί. Ήδη έχουν εκπαιδευτεί 7, ε, 7 μεραρχίες. Άλλη περίπτωση. υπάρχει κρίση, δεν στέλνουμε αποστολή, αλλά θέλουμε να ενισχύσουμε τον τόπιο δυναμικό των χωρών. Χωρίς να μπούμε συγκεκριμένο παράδειγμα, ας δούμε τι γίνεται στο μέλλον. Αυτό κάνουμε. Βλέπουμε τον χώρο που κινείται η ISIL ή η ISIS. Και μία από τις προκλήσεις ποια θα είναι, να ενισχύσουμε τις χώρες της περιοχής. ούτω ώστε οι χώρες να έχουν τη δυνατότητα να είναι πιο ανθεκτικές. Διότι εάν καταφέρουμε να νικήσουμε αυτή τη μάστιγα που αποκαλείται ISIS. Αν δεν γεμίσουμε το κενό και αν δεν ενισχύσουμε τις χώρες της περιοχής, πάντα κάποιος θα εμφανίζεται. Κάποια άλλη ε, τρομοκρατική ομάδα. Σαν το νερό που γεμίζει τα κενά. Άρα πρέπει να ενισχύουμε τις χώρες της περιοχής για να μην εντοπίζουμε το ίδιο πρόβλημα ξανά σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Και το τρίτο, πρόληψη των κρίσεων. Ανέφερα την Αφρικανική Ένωση η ενίσχυση της αεροπορικής δυνατότητας διαχείρισης κρίσεων, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Γιατί δεν ισχύει ότι φτιάχνουμε τέτοιου είδου δυνατότητες για καιρό πολέμου, αλλά τις φτιάχνουμε ή εν καιρό πολέμου, τις φτιάχνουμε εν καιρό ειρήνης. Άρα δηλαδή εκεί το παιχνίδι είναι λιγάκι διαφορετικό. Αυτά είχα να πω. Ε, για την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό. Επίσης ε, προσπαθούμε να στήσουμε και κάποια πιλωτικά σκηνικά ε, και ελπίζουμε να πάρουμε τον Νοέμβρη την εντολή από τους υπουργούς και να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στο Μαλί ή στη Σομαλία συγκεκριμένα. Τώρα, θα ήθελα να αναφερθώ στην ολιστική προσέγγιση. γιατί με μια ολιστική προσέγγιση η διαχείριση κρίσης από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αποτελεσματική και προσφέρεται η δυνατότητα αποτελεσματικής αντίρρησης. Αυτό σημαίνει ολιστική προσέγγιση. Δηλαδή χρήση μιας πολύ μεγάλης εργαλειοθήκης ξεκινώντας από τη διπλωματία, φτάνοντας στην αναπτυξιακή βοήθεια, στο εμπόριο μέχρι και στα στρατιωτικά μέσα. Αυτή η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει τα πάντα. Όλα αυτά τα εργαλεία που διαθέτουμε. Και θα αναφέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Στο κέρας της Αφρικής η επιχείρηση Αταλάντα που είναι μια επιχείρηση για την αντιμετώπιση της πειρατείας και το ΝΑΤΟ έχει τη δική του την αποστολή. Η διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι η προσπάθεια του ΝΑΤΟ ε, ασχολείται μόνο με το σύμπτωμα του προβλήματος, δηλαδή καταδιώκει τους πειρατές και προσπαθεί να εξασφαλίσει το ΝΑΤΟ ότι δεν θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα. Ενώ η προσέγγιση Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαφορετική γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αντιμετωπίσει και τις ε, ρίζες ε, της πειρατείας στην ξηρά. Και εδώ και δύο χρόνια πρέπει να σας πω δεν υπήρξε ούτε μία επιτυχημένη επίθεση, πειρατική επίθεση στην περιοχή. Άρα δηλαδή θα μπορούσε κανείς συμπεράνει, πολύ ωραία, τα καταφέραμε, ας επιστρέψουμε στα σπίτια μας και τέλος ε, έκλεισε η επιχείρηση Αταλάντα. Όμως είμαστε άραγε σίγουροι <clears throat> ότι τη στιγμή που θα αποσύρουμε τα σκάφη μας δεν θα ξαναεμφανιστεί η πειρατεία. Προφανώς και θα ξαναεμφανιστεί γιατί ακόμα δεν έχουμε κατορθώσει να αντιμετωπίσουμε τα αίτια γιατί προέκυψε ε, το φαινόμενο της ε, πειρατείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει μέσα από διάφορους ε, τρόπους. Έχουμε μία δυνατότητα είναι ε, στρατιωτικής εκπαίδευσης. Μετά προσφέρουμε διάφορες δυνατότητες στην αστυνομία, ε, στο στρατό. Ε, επενδύουμε εκεί πάρα πολλά χρήματα. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί σωστά ένα πρόβλημα. Αυτά όσον αφορά την ολιστική προσέγγιση. Το μαλλί, και αυτό είναι άλλο ένα πείραμα, αν μου επιτρέπετε να το χαρακτηρίσω έτσι, Δηλαδή προσπαθούμε και εκεί να εφαρμόσουμε ένα συνδυασμό των που διαθέτουμε. Θα πω τώρα και λίγα λόγια. Γι' αυτό ε, που αναφέρεται στα συμπεράσματα του Δεκεμβρίου του Συμβουλίου όπου δίδεται εντολή στην ύπατη εκπρόσωπο να αξιολογήσει το διεθνές περιβάλλον σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι μια συμβαστική λύση από αυτό που είχε ε, αναζητηθεί αρχικά, δηλαδή μια νέα στρατηγική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, τι μορφή θα λάβει αυτή η στρατηγική, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Ακούσαμε και το είπε ε, και εδώ στο Κοινοβούλιο η ύπατη εκπρόσωπος ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στο να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα μεγάλα θέματα. Αλλά ξέρετε ούτε και αυτή γνωρίζει αυτή τη στιγμή ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να ε, καταλήξουμε σε μία σωστή στρατηγική. Εδώ θα σας αναφέρω την καθαρά προσωπική μου άποψη που βέβαια βασίζεται σε μία εμπειρία πέντε μηνών και παρόλα αυτά ξεκολουθώ να έχω την οπτική γωνία του εξωτερικού παρατηρητή να πω το εξής ότι όσον αφορά την στρατική ασφάλειας ε, που εξακολουθεί να ισχύει θεσπίστηκε το 2003 μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο περιβάλλον και για πολύ συγκεκριμένους στόχους. Στόχος ήταν να βοηθήσουμε ε, στο να συμφιλειωθεί αυτή η βαθιά διχασμένη κοινωνία του Ιράκ. Ε, αυτή η στρατηγική ήταν θαυμάσια, δεν υπάρχει αμφιβολία από αυτού, όμως αν δείτε λιγάκι το πώς ξεκινάει όλη η στρατηγική, ξεκινάει με τα εξή λόγια. Η Ευρώπη δεν ήταν ποτέ τόσο ελεύθερη, τόσο ασφαλής ε, και τόσο ευημερούσα. Είναι λοιπόν αυτή η στρατηγική ε, που εκφράζει την τρέχουσα άποψή μας, δεν είμαι σίγουρος από αυτού κυρίως όσον αφορά στις ε, δύο μεγάλες προκλήσεις ε, που προέκυψαν κατά τα τελευταία έτη ε, ή κατά το τελευταίο καιρό μετά από την προσάρτηση της Ουκρανίας στη Ρωσία και μετά από την ταχύτατη επέκταση του Ισλαμικού κράτους, του Άσις. Και κάτι άλλο, μετά από αυτά που βιώσαμε στην Ανατολική Ευρώπη. Ποια είναι η σχέση μας με τη Ρωσία. Κάτι θα έπρεπε να πούμε από αυτού και για την τρέχουσα κρίση αλλά και για το μέλλον. Πώς τα βλέπουμε όλα αυτά. Αυτό είναι ένα καθαρά στρατηγικό θέμα. Δεν έχουμε απαντήσει ακόμα στην αλλαγή που γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. αυτό το σημείο επαφής ε, ανάμεσα στην ε, μεγαλύτερη ε, και την μικρότερη γειτονία Αν δείτε λοιπόν τις εθνικές ε, στρατηγικές ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαπιστώσετε ότι όλες ε, συμπεριλαμβάνουν πρώτα απ' όλα τις κυβερνοαπειλές. Οι κυβερνοαπειλές υπάρχουν δεν αντιμετωπίζονται στην στρατηγική μας ασφαλείας. Άρα δηλαδή είναι απαραίτητο να υπάρξει κάποια επικαιροποίηση και λόγω αυτού και επιπρόσθετα είναι απαραίτητο να ορίσουμε τις προτεραιότητές μας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Έχει φτάσει η στιγμή να είμαστε λίγο πιο σαφείς. Αντί να μας παρασύρουν τα γεγονότα, να είμαστε λιγάκι πιο συγκεκριμένοι και να μην ε, αντιδρούμε, να περιμένουμε να αντιδράσουμε στα γεγονότα εκ των υστέρων, να έχουμε μόνοι μας μια στρατηγική, ένα όραμα. Και κατόπιν τούτου να δημιουργήσουμε μια ισορροπία ανάμεσα στις φιλοδοξίες μας, στο ύψος των φιλοδοξιών μας και τους πόρους που διαθέτουμε. Και θα επανέλθω σε αυτό αργότερα. Γιατί αυτή η ισορροπία δεν υπάρχει ή, εν πάση περιπτώσει, και αν υπάρχει, πολύ αμφισβητούν κατά πόσον έχουμε τους απαραίτητους πόρους για να καλύψουμε τις φιλοδοξίες μας. Και όσον αφορά και τις εταιρικέ σχέσεις, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, με χώρες αλλά και με οργανισμούς όπως είναι το ΝΑΤΟ. Επίσης ε, ε, είδαμε ότι στην Ουαλία πρόσφατα το ΝΑΤΟ ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετάσχει γιατί από μόνο του δεν μπορεί να τα απεξέλθει, δεν θέλει να τα Όσον αφορά λοιπόν τη διαχείριση των κρίσεων και τις επιχειρήσεις που αναπτύσσονται, θα γνωρίζετε ότι έχουμε συνολικά αναπτύξει 17 επιχειρήσεις. 7 εξ αυτών είναι καθαρά στρατιωτικές, οι υπόλοιπες ε, πολιτικές. Συνολικά απασχολούμε στις 17 ε, αποστολές και επιχειρήσεις 7.000 άτομα που δεν είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Και μόνο φέτος δρομολογήσαμε τρεις νέες αποστολές. Η μία είναι στην Ουκρανία, είναι μεταρρύθμιση του τομέα ασφαλείας και παροχής βοήθειας. Μία άλλη είναι η CAR, στην Κεντρική Αφρική. Είναι μια στρατιωτική επιχείρηση γεφύρωσης αν θέλετε και η ΟΚΑΠ ε, στο Μαλί ε, και από ό,τι φαίνεται και από τον τίτλο αυτής της αποστολής είναι το να δημιουργήσει την υποδομή, της ε, ικανότητες να γίνει κάτι. Αυτά από το 2003. Από τότε έχουμε συνολικά αναπτύξει 13 αποστολές και επιχειρήσεις. Και αναφέρω αυτό τον αριθμό για να σας πω μεταξύ άλλων ότι κατορθώσαμε και ορισμένες εξ αυτών να τις ολοκληρώσουμε. Όχι δηλαδή να τις ε, συστήσει κανείς και μετά να παραμένουν στο διήνεκες. Εμείς κατορθώσαμε κάποιες εξ αυτών να τις ολοκληρώσουμε κάτι που κατά την άποψή μου είναι χρήσιμο. Ε, αποδίδεται μεγαλύτερη έμφαση τόσο στο στρατιωτικό όσο και στο πολιτικό σκέλος. Μεταρρύθμιση ε, της ασφάλειας, ε, εκπαίδευση ε, σε θέματα στρατιωτικά αυξάνεται η παροχή βοήθειας σε αυτόν τον τομέα. Κάτι άλλο το οποίο ήδη ανέφερα. Ε, καμία από αυτές τις αποστολές δεν είναι βραχυπρόθεσμη ή βραχύβια. Σπάνια υπάρχει αυτό. Πολλοί πιστεύουν ότι τα εργαλεία της Κομισιόν ε, είναι όλα μακροπρόθεσμα ενώ η, ε, τα εργαλεία της ΚΠΑ είναι όλα βραχίδια. Θα δω τώρα, θα δούμε δύο αποστολές που ξεκίνησαν φέτος. Η μία είναι Ουκρανία, η άλλη είναι ε, κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία. Η μία είναι στρατιωτική, η άλλη πολιτική. Πάρουμε, ας πάρουμε την Ουκρανία. Εκεί η αποστολή υποτίθεται έχει ε, την διάρκεια ζωής ε, για δύο χρόνια για να επανέλθει η ασφάλεια στην Ουκρανία με μια στρατηγική αναθεώρηση ήδη μετά την πρώτη χρονιά. Και μίλησα σε ένα συνάδελφο που είπε ότι δίρκεσε η ε, αποστολή για 15 χρόνια. Κοιτάξτε, αυτά όλα είναι για δύο χρόνια. Αν όμω θέλει κανεί να τα κάνει πιο σωστά, διαρκεί πολύ περισσότερο. Η αποστολή CAR ξεκινήσαμε ε, ε, ως στρατιωτική αποστολή EU4RCA και μέχρι να φτάσουν ε, τα στρατεύματα των ΗΕ Μινούσκα. Πάντως, όταν παραδίδαμε το κουμπί στη Μινούσκα θα μπορούσε κανείς να πει ότι μπορούσαμε και να φύγουμε. Όχι, αυτό δεν ισχύει. Δεν θα πρέπει ούτε μία στιγμή να σκεφτόμαστε ότι όταν παραδίδουμε το κουμπί ότι μετά ε, αποφασίζουμε αν θα παραμείνουμε όχι στη χώρα. Όχι, η απόφαση λαμβάνεται εκ των προτέρων. Και αν δεν θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά με μισή καρδιά και να αποτυγχάνουμε, τότε πρέπει να παραμένουμε στη χώρα. Και αυτό είναι ένα κομμάτι της δουλειάς μας. Βέβαια αυτό δεν το ανέφερα, όμως υπάρχουν αυτές οι στρατηγικές ε, μετάβασεις, δηλαδή πώς μετακινούμεθα ανάμεσα στα διάφορα εργαλεία. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να τα βλέπουμε όλα αυτά ε, μέσα στην πολυπλοκότητά τους ε, με τον τρόπο αυτό ε, διοργανώνουμε τις επιχειρήσεις μας και τις αποστολές μας. Και οι αποστολές ε, αυτές ε, είναι ένα κομμάτι πολλών περισσότερων. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα που αφορά στη χρηματοδότηση σε σχέση με τα διλήμματα που υφίστανται. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Και Νομίζω ότι ε, στην ε, πολιτική ασφαλείας κατά τους επόμενους μήνες ε, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα να δούμε μία προς μία τις αποστολές για να δούμε κατά πόσον κάποια μπορεί να ολοκληρωθεί, αν μπορούμε να έχουμε επιπρόσθετες επιπρόσθετη εξοικονόμηση κονδυλίων, γιατί δεν υπάρχουν πια χρήματα στον προβλησμό. Δεν μπορούμε να αναπτύξουμε άλλη επιχείρηση. Αν, ας πούμε, ε, μας επιτρέψουν οι συνθήκες να αναπτύξουμε μία αποστολή ειρήνη στη Γάζα, δεν υπάρχουν χρήματα. Ωραία τα λέμε, αλλά στον προπολογισμό δεν προβλέπεται ούτε ένα ευρώ, τίποτα. Άρα δηλαδή πρέπει να δούμε ποια επιχείρηση θα πρέπει να κριθεί ολοκληρωθήσα για να κάνουμε εξοικονόμηση κονδύλιων όπως σας είπα. Και πάλι αυτά που θα πω, πω αφορούν ε, τον εσωτερικό τρόπο των δικών μας σκέψη. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ να μην καταλήξει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Μία από τις μεγαλύτερες ε, πολιτικές αποστολές είναι στη Γεωργία η οποία ξεκίνησε για να ε, βοηθήσει να εφαρμοστεί η συμφωνία του 2008. Εκεί έχουν εγκατασταθεί 283 άνθρωποι. Το θέμα που τίθεται είναι κατά πόσο τους χρειαζόμαστε όλους αυτούς. Καθαρά πολιτικά θα μπορούσε καλής ε, να ισχυριστεί ότι ήταν ανόητο, λάθος, ε, θα εξέπεμπε πολύ κακό μήνυμα τώρα προς τη Ρωσία, αν μειώναμε τον αριθμό αυτών των ανθρώπων. Θα προέβαιναν σε παρερμηνία. Και υπάρχει μόνο μία λύση. Αν δεν υπάρξει αναδιάρθρωση της βοήθειάς μας προς τη Γεωργία που πρέπει να το κάνουμε διότι η χώρα έχει συνάψει συμφωνία σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε πιο αποτελεσματικά και αν μπορούμε να έχουμε ένα πακέτο το οποίο αναδιοργανώνει όλα αυτά τα εργαλεία και γινόμαστε πιο αποτελεσματικοί, γιατί να μην το κάνουμε. Όμως όλα αυτά τα ερωτήματα είναι ανοιχτά. Εγώ απλά θίγω κάποια θέματα. Ορισμένα εξ αυτών των θεμάτων αποτελούν διλήμματα. Δεν έχουμε συμφωνήσει από αυτών και θα ήθελα απλά να τα συνειδητοποιήσετε όλα αυτά γιατί εμάς μας ενδιαφέρει να συμμετέχουν σε αυτές, συμμετέχει σε αυτές τις και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τώρα τις εταιρικές συνεργασίες και συμφωνίες Υπάρχει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον ε, από πλευρά των εταίρων μας, των χωρών και των οργανώσεων θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας και ορισμένοι εξ αυτών άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι απλή οικονομική ένωση, είναι πολύ περισσότερο από αυτό. Έχει εξωτερική πολιτική, έχει πολιτική ε, ασφάλειας και άμυνας, έχει τη σχετική υποδομή. Ας ξεκινήσουμε με τους διεθνείς οργανισμούς. Ε, προφανώς τα Ηνωμένα Έθνη είναι το πλαίσιο, η ομπρέλα που καλύπτει τα πάντα. Ό,τι και να κάνουμε στον τομέα αυτό θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με το διεθνές δίκαιο το οποίο πρεσβεύουν τα Ηνωμένα Έθνη. Συνεργαζόμαστε με τα Ηνωμένα Έθνη σε θέατρα πολέμου, στο Μαλί, στο Αφγανιστάν, ε, σε όλα αυτά τα σημεία. Υπάρχει μια πολύ στενή σχέση. Επίσης έχουμε και διάλογο υψηλού επίπεδου με τη μορφή μιας υψηλής συγκεκριμένης ομάδας ε, ε, συνεργασίες με το Ηνωμένα Έθνη συγκρίνουμε τι σημειώσει μα ε, και κάθε εβδομάδα μιλάμε με τους συναδέλφου μα στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτή είναι μία ε, σχέση εργασίας. Όσον αφορά τώρα το ΝΑΤΟ, ε, πολλές φορές από το ΝΑΤΟ αντλούμε απογοήτευση γιατί βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε πάνω από ένα επίπεδο. Από την άλλη πλευρά, κάτω από τα ραντάρ Όσον αφορά την πρακτική συνεργασία, ήδη γίνονται πάρα πολλά. Αλλά όμως υπολείπονται ακόμα πάρα πολλά και πρέπει να γίνουν. Και νομίζω ότι είμαστε αποφασισμένοι να εντοπίσουμε αυτούς τους τονείς όπου υπολείπονται πάρα πολλά για τη συνεργασία μας με τον Άτομο. Ένα παράδειγμα είναι αυτός ο υβριδικός τρόπος πολέμου που βγαίνει, απορρέει σαν πρόταση από το Συμβούλιο. Το ΝΑΤΟ περιμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απλώς εργαλεία στα χέρια των κρατών μελών. Και δεν θα σε εκπλήσει ότι τα κράτη-μέλη θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν όλα τα εργαλεία στη διάθεσή τους ε, αποτελεσματικότερα. Και θα σε εκπλήσει αυτό που σας λέω. Αυτός είναι ο βασικός άξονας αν θέλετε. Δεν ανέφερα την επόμενη σύνοδο κορυφής του Ιουνίου του 2015 που θα συζητήσει τα θέματα ασφαλείας και άμυνας. Και θα πρέπει να πούμε πού βρισκόμαστε όσον αφορά τα 60 καθήκοντα που μας ανέθεσαν. θα πρέπει να εντοπίσουμε και νέους τομείς ασφαλείας και άμυνας συνέχεια να συζητούμε ε, την άμυνα και μετά τον Ιούνιο του 2015. Και άλλο στοιχείο. Θα, θα πρέπει να ανταποκριθούμε και στα όσα εκφράστηκαν στην Ουαλία. Ανάμεσα ε, ε, στις δύο συνόδους κορυφής, η σύνοδος της Ουαλίας μπορεί να θεωρηθεί ένα ενδιάμεσο γεγονός. Απευθύνθηκαν σαφείς εκκλήσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί να βοηθήσει σε διάφορους τομείς. Οι χώρες εταίροι. Έχουμε 16 χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνίες πλαίσια συμμετοχής με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ χρήσιμο πρακτικό εργαλείο. Μπορούν χωρίς να περάσουν από εμπόδια οικονομικά και άλλα να μπορούν να στείλουν κάποιον να συνεργαστεί, να εργαστεί στις αποστολές μας. Είναι ένα εργαλείο που φροντίζει αυτό το πρόβλημα για όλους εκείνους που έχουν υπογράψει. Είναι ένα πρακτικό εργαλείο αλλά και σημαντικό πολιτικό μήνυμα στέλνει ότι χώρες δηλαδή από την Ασία συμπεριλαμβανομένες της Νότια Κορέας, της Αυστραλίας, της Λατινικής Αμερικής είναι χώρες που θέλουν να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπογείως ε, έχουμε πολλούς εταίρους. Η Αταλάντη έχει γίνει ε, πολύ ενδιαφέρον, ενδιαφέρουσα βάση για κάτι τέτοιο. Έχουμε η Ιαπωνία, Κίνα, Κολομβία που συνεργάζονται που θα συμβάλλουν με πλοίο στις ε, επιχειρήσεις κατά των πειρατών. Και τέλος κάποια διλήμματα στα γρήγορα. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα, τις μεγάλες προκλήσεις όπου χρειαζόμαστε και πολύ μάλιστα την υποστήριξή σας την επόμενη περίοδο είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι πτυχές ασφάλειας και άμυνας θα συμπεριλαμβάνονται στον ευρύτερο προβληματισμό και δράση της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Αλλά είναι κρισίμου σημασία. Επειδή η άμυνα σε πολλές, από πολλές πλευρέ θεωρείται ότι είναι κάτι κακό, σε πολλού χώρου θεωρείται κάτι κακό. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να συνεχιστεί, δεν είναι βιώσιμο. Μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε μια σφαιρική, μια ολιστική προσέγγιση. Άλλο δίλημα. Οι 17 αποστολέ και επιχειρήσει. Κάποιοι έθεσαν ερωτήσει. Είπαν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μπορούμε να καταφέρουμε τόσε πολλέ. Βέβαια αυτό πάντα εξαρτάται από την υποστήριξη που παρέχουμε. Από πλευράς στελεχών, στελέχωσης μπορούμε. Το πρόβλημα που έγκυται στην ισορροπία μεταξύ φιλοδοξιών και πόρων. Εάν δεν αλλάξουμε την ισορροπία, δεν γίνεται κάτι. Να λέμε ότι έχουμε 17 αποστολές και επιχειρήσεις. Και το μεγαλύτερο τμήμα του προπολογισμού της ΚΕΠΑ ε, καταναλώνεται για την υποστήριξη των πολιτικών αποστολών και αν πούμε ότι έχουμε 260 εκατομμύρια διαθέσιμα. Δεν είναι μεγάλο ποσό. Ξέρουμε όμως ότι δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε μόνο περιορισμένους πόρους. Αυτή ήταν η συμφωνία μεταξύ κρατών μελών. Το μήνυμά μου είναι το εξής. Χρειάζεται ισορροπία αν έχουμε μικρότερο ποσό για να υποστηρίξουμε τέτοιου είδους δραστηριότητες άμυνας πρέπει να μειώσουμε τις φιλοδοξίες. Αν έχουμε αυτού του επίπεδου τις φιλοδοξίες και το διατηρήσουμε το επίπεδο, τότε πιθανότατα θα πρέπει να αυξήσουμε τους πόρους. Άλλο δίλημα. ταχεία ανταπόκριση, ταχεία αντίδραση. Ε, είναι πολύ κρισίμου σημασία. Στο ΝΑΤΟ ε, έχουν εστιάσει τις προσπάθειες τους αλλά αφορά συλλογική άμυνα, αλλά και για την διαχείριση των κρίσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε εργαλεία που είναι άμεσα διαθέσιμα και μπορούμε να τα αναπτύξουμε, να τα συντηρήσουμε και να τα προωθήσουμε γρήγορα. Έχουμε ένα υπέροχο εργαλείο. Τις ε, μονάδες μάχης, battle groups είναι πολύ καλή, καλό μέσο. Αν το συγκρίνουμε με το ΝΑΤΟ, το RNF, δηλαδή τη δύναμη αντίδρασης του ΝΑΤΟ, από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι διαθέσιμο η μονάδα εντός δεκαημέρου 30 μέρες στο ΝΑΤΟ. Πριν την μεταρρύθμιση, λέει η Πρόεδρος, συμφωνεί και ο μιλητής, ναι, ε, βλέποντας τι αυτά που είδαμε όλοι μας, τι κάνανε οι Ρώσοι, οι 30 μέρες ε, ανήκουν στην ιστορία πια. Είναι πάρα πολύ μεγάλη χρονική περίοδος. Αλλά αυτή η μάχημη μονάδα ε, ε, είναι κάτι υπέροχο, αλλά δεν έχει αναπτυχθεί, δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα και δεν έχει αποδείξει ακόμα πόσο αξίζει το Battle Group. Το πρόβλημα δεν είναι το όλο οικοδόμημα η δυνατότητα που υπάρχει, αλλά η πολιτική βούληση είναι πολιτικό το πρόβλημα και αυτό είναι κάτι για το οποίο χρειαζόμαστε πολύ την υποστήριξή σας. Να έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα ξεπεραστούν οι δυσκολίες. Εν μέρη τα προβλήματα αφήνονται στην ε, χρηματοδότηση, εν μέρη στις ε, λήψεις αποφάσεων, αλλά και τα δύο είναι πολιτικής χρειάς ζητήματα. οι χώρες θέλουν να αναπτύξουν δυνάμεις σε κάποια περιοχή και δεν ταυτίζεται ε, με τους άλλους που θέλουν ένα γενικό πλαίσιο για να υπάρχει δύναμη σε τιμότητα κλπ. Η χρηματοδότηση είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, πολύ μεγάλο. Αν συνεχίσουμε να περιμένουμε χώρες που δεν έχουν συμφέρον σε κάποια περιοχή να διακινδυνεύσουν τις ζωές των στρατευμάτων τους και να χρηματοδοτήσουν την αποστολή, δεν πάμε πουθενά σε περίπτωση κρίσης. Ποιος πολιτικός θα γυρίσει στην πατρίδα του και θα εξηγήσει στο εκλογικό του σώμα ότι πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ δύσκολο. Θα πρέπει ίσως να αλλάξουν οι κανόνες. Το ίδιο και για το pooling και sharing, δηλαδή τον, τη συλλογή της συνάρτησης των δυνάμεων και τον καταμερισμό των ευθυνών ε, και των δυνάμεων. Είναι σημαντικά αυτά σαν στόχοι που έχουν δρομολογηθεί. Παραπέμπω ξανά στο Δεκέμβριο του 2013 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα μη επανδρομένα επτάμενα σκάφη, τα drones. Ένα αέριο ανεφοδιασμός αεροσκαφών. Υπάρχουν μεγάλα κενά. Και ελπίζουμε ότι θα πρέπει να δοθούν αυτές οι δυνατότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ καλές δυνατότητες αυτές. Αλλά το θεμελιώδες πρόβλημα και το ίδιο ισχύει για το ΝΑΤΟ με την ευφύ άμυνα. Εάν δεν αντιμετωπιστούν βασικά προβλήματα σωστά, κυρίως η διαθεσιμότητα, διαθεσιμότητα των ικανοτήτων, αν δεν αναπτυχθούν, αναπτυχθεί δυνατότητα, αν δημιουργούνται ικανότητες, δηλαδή μια χώρα να ξέρει ότι μπορώ να βασιστώ σε συγκεκριμένες ικανότητες και δυνατότητες, δεν θα αλλάξει η αντίληψη που υπάρχει όσον αφορά τις αντιλήψεις μας και θα εξακολουθεί να υπάρχει αλληλεπικάλυψη προσπαθειών. Τέλος. Στήριξα την νέα στρατηγική, εκτενώς, όπως θα καταλάβατε από αυτά που λέω. Απ' την άλλη πλευρά, γνωρίζω ότι υπάρχουν και αντεπιχειρήματα. Και ένα από τα μεγαλύτερα είναι ότι άμα, άμα ξεκινάς κάτι δεν ξέρεις μετά αν μπορεί να το διορθώσεις. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ κρατών μελών και υπάρχουν κρίσιμα στατικικά ζητήματα μεταξύ χώρων μελών. Ποια είναι η απάντησή μου σε αυτό. Από τη μία πλευρά είναι σημαντική η διαδικασία, να συζητούμε δηλαδή στατικικά ζητήματα. Είναι σημαντικό, συζητούμε προτεραιότητες, πώς να αντιδρούμε σε κάποιες νέες εξελίξεις. Και Εάν οι διαιρέσεις είναι τόσο βαθιές, οι τόσο βαθιές, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι αν κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί ή αν δεν τα κουβεντιάζουμε είναι η σωστή προσέγγιση. Θα σταματήσω εδώ. Συγγνώμη που υπήρξα τόσο εκτενής και είμαι ακόμα στο στάδιο της εισαγωγής αλλά υπάρχουν τόσα πολλά βλέπετε που πρέπει να κουβεντιάσουμε και πραγματικά χρειαζόμαστε σας, την υποστήριξή σας, την πολιτική σας υποστήριξη και να καταλάβουμε και εμείς ποιες είναι οι δικές σας σκέψεις και απόψεις για να τις λάβουμε υπόψη στο δικό μας προβληματισμό. Εκτιμώ πάρα πολύ τη δυνατότητα που μου δώσατε να μιλήσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, πριν λοιπόν ε, δώσω το λόγο στα μέλη της Επιτροπής, ε, για να σας υποβάλω ερωτήσεις κύριε Ικλόντι, θα ήθελα να πω το εξής. Τη Δευτέρα είχαμε μία συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων η οποία ασχολήθηκε αποκλειστικά και μόνο με την κατάσταση στη EULEX στην αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο Κωσυφοπέδιο. Πολύ ψηλό επίπεδο υποτίθεται και γι' αυτό η κατάσταση είναι πάρα πολύ λεπτή, ευαίσθητη. Οφείλουμε ε, ταχύτατα να εξετάσουμε αυτό το πρόβλημα και με σοφό τρόπο. αποφασίσαμε να έχουμε το συντομότερο δυνατόν και την αντίληψη της ύπατης εκπροσώπου. και τα μέλη πιστεύουν ότι θα πρέπει να ε, υπάρχει μηδενική ανοχή αν τελικά αποδειχθεί ότι ευσταθούν κάποιες ε, αιτιάσεις, ε, κάποιες υπόνοιες Τώρα λοιπόν έχουμε τις αντιδράσεις ε, των ε, μέσων ενημέρωση, αλλά και των στελεχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορώ λοιπόν να σας ε, υποσχεθώ ότι θα υπάρξει μία συνεδρίαση του Διευρυμένου Προεδρίου της ΣΕΝΤΕ και κλεισμένων των θυρών και κατόπιν θα συντονιστούμε με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και θα πρέπει να εξετάσουμε ειδικά θέματα ασφάλειας και άμυνας. Η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη καθότι όλη αυτή η έννοια της ΚΠΑ έχει άμεση σχέση με την κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια. Γι' αυτό λοιπόν όλα αυτά δημιουργούν κάποιες δυσκολίες. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Γκόμεσε, στην Άννα Γκόμεσε. Παρακαλώ κυρία Γκόμεσε. Ευχαριστώ ε, κυρία Πρόεδρε. Ε, ευχαριστούμε κύριε Ικλόντι. Και πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ, όχι μόνο όλο το υποβαθρό σας για να αντιμετωπίσετε τις προσκλήσεις που υπάρχουν, αλλά μου άρεσε και η παρέμβασή σας που έδειξε ότι έχετε κατανοήσει τις μεγάλες προκλήσεις που υπάρχουν. Λυπάμαι που είμαστε τόσοι λίγοι εδώ σήμερα, γιατί νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να υπάρχουν περισσότεροι. Αλλά από ό,τι φαίνεται η συνάδελφοί μου ε, έπρεπε να πάνε κάπου αλλού. Είμαι σίγουρη ότι θα βρεθούν και άλλες ευκαιρίες για να ξανασυζητήσουμε. Πάντως μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η γενική επισκόπηση που παρουσιάσατε και το ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν ε, στρατηγικής φύσεως ε, σκέψεις για όλα αυτά που κάνουμε. Μου άρεσε το ότι αποδώσετε ιδιαίτερη σημασία στο οικονομικό στοιχείο και επίση μου άρεσε και το ότι καλείται όλους να προσαρμοστούν στις νέες προκλήσεις. Το μόνο με το οποίο διαφωνώ είναι αυτά που είπατε για τη Λιβύη. Γιατί εγώ τα τελευταία χρόνια έχω παρακολουθήσει από, κοντά ε, την κατάσταση στη Λιβύη. Ήμουν εισηγήτρια του Κοινοβουλίου το 2010 και την έχω επισκεφτεί επανειλημμένα. Ξέρετε στη Λιβύη δεν ήταν ε, ότι δεν υπήρχαν δυνατότητες να παρέμβουμε. Αυτά που δίδαμε στον Καντάφη τα δίδαμε και στους επόμενους, κυρίως έχοντας κατά νου ότι στη χώρα αυτή το μόνο που δεν έλειπε ήταν τα χρήματα. Πάντως ε, το 2012 πήγαμε με το Κοινοβούλιο με μια αποστολή της Επιτροπής ε, Εξωτερικών Υποθέσεων. Ο κύριος Ντανζόν ήταν τότε πρόεδρος της Υποπιτροπής και αυτό που είδαμε και είπαμε επανειλημμένα είναι ότι χρειαζόμαστε μια στρατηγική πολιτική για τη Λιβύη Μιλάμε, δεν είναι ένας τυχαίος γείτονας, ένας γείτονας που είναι μόνο μια ώρα από τις ακτές μας, με πολλά όπλα, πολλά χρήματα και ένα πλήρες κενό θεσμικό. Αν λοιπόν ήρθαν κάποιοι να μας επισημάνουν τι δεν κατορθώσαμε να επιτύχουμε, προφανώς αυτό που μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να συστήσει θεσμούς, δεν έγινε ποτέ όμως κάτι τέτοιο. Και αυτό ήταν λάθος των Ηνωμένων Εθνών, γιατί θυμάμαι πάρα πολύ καλά ε, τις μεγάλες συζητήσεις που είχαμε τότε με τον εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών. Θυμάμαι και τις συζητήσεις με τα κράτη-μέλη και θυμάμαι και ότι είχαμε μία ύπατη εκπρόσωπο που δεν καταλάβαινε τι διακυβεύεται. Και η Ευρώπη Ήτανε η μόνη που θα μπορούσε, με άλλους βέβαια, να βοηθήσει σε αυτό το κεντρικό θέμα του SSR, DDR. Γιατί τι νόημα έχει να στείλει κανείς μια αποστολή αν δεν υπάρχει ε, ένα υποδομή. Μίλησα με κάποιους ε, που θα πήγαν εκεί ε, και μου είπαν ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν αλλά Κάθε φορά που βρίσκουν κάποιον να συνομιλήσουν, τελικά αυτός μετατίθεται στην έρημο και ξαφνικά χάνεται και η γνώση. Γιατί δεν υπάρχει κεντρική διοίκηση. Ο στρατός και η αστυνομία κατόνομα υπάρχουν. Και αυτό νομίζω ήταν προφανές για όλους που δεν είναι ειδικοί σε θέματα ε, στρατηγικά και ασφαλείς όπως είμαι εγώ. Μπορώ λοιπόν να φανταστώ ότι όλα αυτά συνέβησαν γιατί υπάρχει έλλειψη Ευρώπης και Ευρωπαίων και ορισμένα κρατημέλη φταίνε περισσότερο από άλλα για αυτή την κατάσταση. Γιατί ξέρετε τι έκαναν, βάζουν ε, ε συμβούλους ε, στα Υπουργεία για να έχουν κάτι να παίξουν και με τον τρόπο αυτό όμως παραμελούν το κεντρικό ερώτημα που είναι πώς οικοδομείται ένα κράτος περίπου το ίδιο συνέβη και με το κοσυφοπέδιο. Και πραγματικά δεν ανταποκριθήκαμε στις υποχρώσεις μας. Ολιγορία ήταν το πρόβλημα. Βεβαίως, μερικοί φέρνουν μεγαλύτερη ευθύνη από άλλους. Εγώ δεν λέω ότι δεν φταίνε ε, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ιταλία και ίσως και η Γερμανία. Και τώρα η κατάσταση είναι αυτή που είναι. Και εξακολουθούν να ολιγορούν η Lady, Lady και εκείνη φέρει ευθύνη. Γιατί νομίζω αυτό το έχει πει επανειλημμένα το Κοινοβούλιο. Και όλα τα ψηφίσματα που θεσπίσαμε για τη Λιβύη έχουν συγκεκριμένες παραγράφους για την αποστολή της ΚΠΑ και οι Λίβοι ήρθαν και σε εμά, όπως πήγανε και στο ΝΑΤΟ, για να παρακαλέσουν για τη βοήθειά μας. Και, μας, και εμείς δεν διαπερθήκαμε καθόλου. Να το λοιπόν το μεγάλο πρόβλημα και δεν έχουμε δει ακόμα τα χειρότερα, γιατί είναι Προφανές ότι στην πολιτοφυλακή θα παρισφρήσουν εγκληματικά και τρομοκρατικά στοιχεία. Σας λέω, δεν τα έχουμε δει ακόμα τα χειρότερα της Λιβύης και να δούμε τι θα κάνουν τα κράτη-μέλη. Άρα δηλαδή αυτό που χρειαζόμαστε είναι καθοδήγηση. Και πιστεύω ότι ο ρόλος της νέας ύπατης ε, εκπροσώπου ε, θα είναι καθοριστικός. Ε, περίμενα ότι η κυρία Άστον, επειδή έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία, μια χώρα με μεγάλη ασφάλεια, θα ήταν αποτελεσματική. Όμως η ίδια τελικά είχε μια πολύ αρνητική προσέγγιση στην ΚΠΑ, λόγω ε, της, του, του ιστορικού της, που είναι Βρετανή πίκος, και λόγω και της Βρετανικής κυβέρνησης. Έχουμε λοιπόν από τη μια την Μεγαλουτανία που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για την ΚΠΑ και προφανώς την κατέστρεψε γιατί πίστευε ότι πρόκειται για μια προνομιούχα στέχη με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον ΝΑΤΟ και μέχρι εκεί, αλλά δεν ισχύει αυτό. Και το άλλο πρόβλημα είναι η Γερμανία εντάξει, έχει μια ειρηνιστική προσέγγιση, μπορεί κανείς να την εξηγήσει με ιστορικούς λόγους και μερικές φορές ε, αρνείται. Ξέρετε, είχαμε και κάποιες γελίες συζητήσει ε, για την ΚΠΑ, ποια θα ήταν η εμβέλειά της και διάφορα παρεμφερή. Το θέμα της χρηματοδότησης και αυτό παίζει ρόλο μαζί με τα άλλα. Σήμερα αναφέρθηκε ότι το θέμα της χρηματοδότησης είναι καθοριστική σημασίας και ελπίζω να μπορείτε να ασκήσετε πίεση τουλάχιστον να υπάρχει χρηματοδότηση για κοινέ αποστολές ε, στο πλαίσιο της ε, ΚΠΑ, της Κοινή Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας. Ε, το σημαντικότερο, όπως σας είπα, η καθοδήγηση και θέλω να πιστεύω ότι η νέα ύπατη εκπρόσωπος θα είναι πιο ευαίσθητη, πιο αποτελεσματική και θέλω να ελπίζω ότι επειδή και η ίδια είναι Ιταλίδα, λόγω αυτού του γεγονότος θα δώσει ιδιαίτερη σημασία στη Λιβύη. Ευχαριστώ κυρία Γκόμες. Um, Επιτρέψτε να θέσω δύο ερωτήσεις. Πολύ σύντομα. Να αναφερθούμε και την, στη Γιούλεξ. Ποια είναι η γενική εικόνα της αποστολής, αναφερθήκατε σε αυτό, θα το συζητήσουμε αυτό και για την κρίση που αντιμετωπίζετε θα συζητηθεί ξεχωριστά. Η ολιστική προσέγγιση είναι η βασική αρχή. Κατά την άποψή σας, τι χρειάζεται για κάθε αποστολή. Και ποια αποστολή θα πρέπει πλέον να αποσυρθεί Δεύτερον, οι ομάδες μάχης, τα battle groups. Πώς το βλέπετε αυτό το θέμα. Το θέμα των μονάδων μάχης. Το επιχειρησιακό τους σχήμα. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε αλληλεπικαλύψεις με την ε, μονάδα ταχείας αντίδρασης, με τις μονάδες ταχείας αντίδρασης του ΝΑΤΟ. Στο ΝΑΤΟ ήδη άρχισε γρήγορα, ε, άρχισε μάλλον ήδη η μεταρρύθμιση της μονάδας ταχείας αντίδρασης. Ποια είναι η άποψή σας σε σχέση με αυτό, σε συνάρτηση με αυτό, ποια είναι η άποψή σας για τις ε, μονάδες αυτές μάχης, τα battle groups. Ε, θα ξεκινήσω με δύο σχόλια. Για τη Λιβύη. Συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό θέλω να πω ότι όλες οι προσπάθειες που γίνονται με στατιωτικά μέσα είναι μακρόπνοες προσπάθειες. Η Λιβύη είναι ζωντανό παράδειγμα. Να μπαίνει κανείς να κάνει κάποιες στατιωτικές επιχειρήσεις και να αποσύρεται. Δεν πετυχαίνεις πολλά έτσι. Χρειάζεται συνεχής προσπάθεια βιώσιμη προσπάθεια. Διαφορετικά η κατάσταση όχι μόνο μπορεί να μην βελτιωθεί αλλά και να επιδεινωθεί. Και για το άλλο θέμα που αναφέρατε, για τα βήματα που ακολουθούμε είναι σημαντικό. Μάθαμε και στο Ιράκ. Δεν αρκεί να μπει κανεί να διαλύσει τις δυνάμεις ασφαλείας και το στρατό και μετά να εκπλήσετε. Ε, που βασιλεύει το χάος στη χώρα μετά. Συμφωνώ. Και ότι η Λιβύη ε, βρίσκεται σε μια περιοχή που είναι σε κατάσταση χαόδη. Ε, ελοχεύουν πολλοί κίνδυνοι. Υπάρχουν πολλές αρνητικές συνέπειες που παραμονεύουν. Για τη χρηματοδότηση της ΚΕΠΑ και των σχετικών αποστολών. Θυμάμαι τον Γάλλο Υπουργό Αμίνη στο Μιλάνο. Είπε κάτι που εξέφραζε το πρόβλημα. Είπε η αλληλεγγύη μας περιορίζεται στο 10%. Αυτό είπε. Αυτό είναι το ποσοστό. Σε μια στατιστική αποστολή χρηματοδοτούμε μέσω του μηχανισμού Αθήνα μόνο το 10% του κόστους. Συμφωνώ. Δεν πρέπει να μας εκπλήσει αν αυτά τα εργαλεία μας δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Τα συμφέροντα δεν αλλάζουν. Τα εθνικά συμφέροντα θα παραμείνουν αυτά που είναι αλλά οι κανόνες χρηματοδότησης είναι κάτι που μπορούμε να αλλάξουμε. Τώρα για τις ε, μονάδες μάχης, τα battle groups. Αν υπάρχει κίνδυνος να επαναλάβουμε κάτι που ήδη γίνεται σε άλλο πλαίσιο. Θα θυμόσαστε ότι Θέλαμε για δύο σκοπούς τις μονάδες μάχης. Πρώτα απ' όλα, ένα εργαλείο μετασχηματισμού το θέλαμε και απ' την άλλη σαν επιχειρησιακό εργαλείο. Σαν μετασχηματικό εργαλείο θέλαμε να βοηθήσουμε τις εθνικές αρχές να μεταμορφώσουν το στρατό τους, να μπορεί να μετακινείται και να αναπτύσσεται πιο εύκολα ανάπτυξη κινητικότητας, εξυγχρονισμός, διαλειτουργικότητα, Σχετικά με αυτό οι μονάδες μάχης σαν έννοια ε, τα πήγαν πολύ καλά. Είναι κάτι που δούλεψε. Το είδα στη χώρα μου, στην Ουγγαρία. Είναι μια καλή έννοια. Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι. Λέμε ότι αυτές οι μονάδες μάχης απέδωσαν όπως έπρεπε και δεν μας νοιάζουν ε, διάφορες άλλες πτυχές. Όχι. Οι άλλες πτυχές δεν είναι ασήμαντες και πόρα απέχουμε από την ολοκλήρωση. Αν επαναλαμβάνουμε προσπάθηση, ή όχι, αν υπάρχει επικάλυψη ή όχι. Μιλάμε τώρα για εθνικές μονάδες που περνούν από εκπαίδευση ε, ε, υπάρχει αξιολόγηση, γίνεται αξιολόγηση μαζί με τον ΝΑΤΟ που εξακριβώνουν ότι οι μονάδες μάχης έχουν τις συγκεκριμένες δυνατότητες που πρέπει. Αυτό είναι καλό. Θα ήταν καλό αν γίνεται. Νομίζω Δεν νομίζω εδώ ότι υπάρχει ένας ιδιαίτερος κίνδυνος, δηλαδή το να καταβάλει κανείς διπλή προσπάθεια το πρόβλημα θα υπήρχε εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση ή αν το ΝΑΤΟ αποφάσιζαν να, κάνουν τα πράγματα συνεργαζόμενοι, αλλά συνήθως συμφωνούν ποιος θα αναλάβει από τους δύο. Α, λοιπόν, είναι διαχειρίσιμο το πρόβλημα. Αν υπάρχει μια κρίση σε μια περιοχή κάπου και μετά περιμένει κανείς και για πολιτικούς λόγους υπάρχει ένα opt-out και λέει όχι επειδή είναι ένας γειτονάς του ας πούμε εάν ε, ε, υπάρχει μια σύγκρουση, υπάρχει ένας μη γραπτός νόμος ε, ότι δεν αναπτύσσει κανείς στρατιωτικές του δυνάμεις στη γειτονική χώρα γιατί καταστρέφονται οι σχέσεις με τους γείτονες και αυτό κρατάει για πολλά πολλά χρόνια. Άρα λοιπόν απέχει κανείς αν δεν, από τη στιγμή που αφορά τη γειτονική χώρα. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει όμως να συνεργάζονται οι δύο, να εναρμονίζουν το έργο τους και να εγγυώνται ώστε θα υπάρχει τουλάχιστον μια δυνατότητα εντάξει μιας κάποιας απόκλησης με ομάδες ε, κατάλληλες ε, κρούσεις, ε, το spearhead κρούσεις όπως το λένε στο ΝΑΤΟ. Έτσι, πάντως είναι διαχειρίσιμο το πρόβλημα, παραλαμβάνω. Για να δούμε. Για τη Βοσνία. Μια επιχείρηση που θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του. Κυρίως επειδή σκεφτόμαστε ότι υπάρχει μία ανάγκη να σεβαστούμε την εντολή και τον ειδικό χαρακτήρα αυτής της εντολής για να μπορέσει κανείς να βοηθήσει. Τα κράτη-μέλη όμως εμφανίζονται διηρημένα στο σημείο αυτό. Και είναι η προσωπική μου άποψη ότι εντάξει η προσπάθεια αξίζει και η επένδυση αυτή και τα χρήματα που έχουμε δαπανίσει τα έχουμε δαπανίσει σωστά, λογικά εάν κάνει κανείς τη σύγκριση με τον κίνδυνο ο οποίος υπάρχει να αποσύρει κανείς τις δυνάμεις και μετά να έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα με τα λέω καιρό, τότε ε, μέχρι και τη Θεσσαλονίκη ξέραμε και τα έχουμε πει και στις ε, Βαλκανικές χώρες ότι καταβάλουμε προσπάθεια, έχουμε αναλάβει αυτή την υποχρέωση, εντάξει, δεν είναι πια ότι εάν θα συμμετάσχουν οι βαλκανικές χώρες, αλλά πότε θα συμμετάσχουν. Και εντάξει, το ξέρω, το καταλαβαίνω και ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο καθένας για την αδυναμία της Βοσνίας να μπορέσει να προχωρήσει, να προοδεύσει σχετικά με τις παραμέτρους οι οποίες και έχουν οριστεί. Και δεν είναι δύσκολες αυτές οι παράμετροι άλλωστε για να τις επιτύχει κανείς δεν ξέρω πόσες φορές επιστρέψαμε, πήγαμε στο Σεράγεβο και τους είπαμε «Μα δεν φοβάστε ότι όλοι οι υπόλοιποι εκεί στην περιοχή σας ε, θα πάρουν το πάνω χέρι και θα ε, πλησιάσουν στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα και εσείς θα μείνετε στην άκρη παραμερισμένοι και εδώ αφορά και το μέλλον σας, τις επενδύσεις σας, το μέλλον, το παιδιό σας. Μην το ξεχνάτε αυτό θα πρέπει να δει κανείς ας πούμε και τις δυνατότητες άμυνας. Αλλά είναι πολύ δύσκολο αυτό το θέμα να λυθεί, δεν νομίζω. Από τη στιγμή που δεν έχει σημασία τότε γιατί ισχύουν αυτές οι παράμετροι. Ακριβώς για να δούμε μπορείτε να παρεμβαίνετε. Ίσως υπάρχει μια παράμετρος που έχει επιλεχθεί λάθος, αλλά να το δούμε ότι το σέβεστε αυτό και μετά να περάσει κανείς την επόμενη φάση και μετά θα βγάλει κανείς ένα συμπέρασμα. Σύμφωνα με την πείρα μου, όσο τη, Βοσ... τη Βοσνία μόνο δεν αφορά μόνο αυτή, αλλά και άλλες χώρες όπως και την Ουκρανία η οποία δεν εφάρμοσε και τόσο καλά όλα αυτά που είχε αναλάβει σαν υποχρεώσεις. για χώρες όπως την Ουγγαρία, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, την ε, Πολωνία, απλά και μόνο να κουνήσει κανείς το καροτάκι και να πει εντάξει πηγαίνετε πίσω και ελάτε ξανά όταν είστε έτοιμοι. Και λειτουργήσε, αλλά στα Δυτικά Βαλκάνια δεν πιάνει αυτό σε όλους και ούτε και στην Ουκρανία επίσης ε, ισχύει. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Εγώ άκουσα πολλές φορές να λένε ότι στα πλαίσια ακριβώς της Ουκρανίας ε, τι θέλουμε. Οι κάτοικοι εκεί να είναι οδηγοί στην όλη διαδικασία. Αυτό όμω είναι λάθος. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι σίγουρα βέβαια είναι κύριοι του εαυτού τους. Θα πρέπει όμως και κάτι να κάνει κανείς για να κερδίσει την ανεξαρτησία του, την αυτονομία του και επίσης και για την ασφάλεια, όλη αυτή τη μεταρρύθμιση πρέπει να είμαστε εκεί επί τόπου και να τους κρατάμε από το χεράκι και να είμαστε σίγουροι πια ότι έκαναν αυτό που έχουν λάβει την υποχρέωση να κάνουν. Θα πρέπει να αλλάξουμε στάση. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να διατηρούμε την ίδια στάση με τις χώρες αυτές όπως το κάναμε στο παρελθόν με άλλες χώρες. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι γίνεται. Ενδιαφερόμαστε να πετύχουμε την Ουκρανία για τις μεταρρυθμίσεις. Ναι, μας ενδιαφέρει, είναι σημαντική αυτή η προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει να τους βοηθήσουμε να πετύχουν όσον αφορά τις αλλαγές τους, τις μεταρρυθμίσεις τους. Αλλά θα πρέπει να τους βοηθήσουμε να είμαστε σίγουροι ότι θα κάνουν τα πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση και τα χρήματα που τους προσφέρουμε, που τους δίνουμε να μην πάνε σε σκοτεινές οδούς, να μην χάνονται. Θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία επίσης. Και αυτό προσπαθούμε, αυτό κάνουμε. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Και Ευχαριστούμε κύριε Κλόντι. Ίσως να κάνω ακόμα, να προβώ σε ένα σχόλιο ακόμα. Τουλάχιστον όσον αφορά την Ουκρανία. Νομίζω ότι αυτά που λέτε είναι λογικά, σωστά τουλάχιστον μέχρι τα Μεϊντάν, μέχρι τα γεγονότα αυτή, γιατί μέχρι τις διαδηλώσεις εκεί, μέχρι τότε η πλειοψηφία της κοινωνίας της Ουκρανίας έδειχνε ότι κρατούσε μια στάση, ότι είχε ένα συγκεκριμένο στόχο και τώρα αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες δυσκολίες όμως, πραγματικές δυσκολίες σε εμπόλεμη κατάσταση. Παρ' όλα αυτά δείχνουν ότι έχουν διάθεση δείχνουν ότι έχουν και διάθεση να ακολουθήσουν τις μεταρρυθμίσεις αλλά να και να το πετύχουν παρόλο τις πολύ δύσκολες συνθήκες. Είναι έτοιμοι να επιφέρουν αλλαγές. Και αυτό και μετά από τις πρόσφατες εκλογές βλέπουμε ακριβώς ότι η κοινωνία τους είναι αποφασισμένο και το έδειξε καθαρά το αποτέλεσμα των εκλογών υπέρ των μεταρρυθμίσεων και υπέρ επίσης της δύση. Μεγαλύτερο μέρος της Ουκρανικής κοινωνίας είναι υπέρ. Αυτό εξέφρασε η πλατεία πλειοψηφία εξέφρασε την άποψη αυτή, τη γνώμη αυτή, την ιδέα αυτή. Τώρα όσον αφορά τη Βοσνία Αρζεγοβίνη. Σίγουρα αυτή η αδυναμία δράσης φαίνεται καθαρά. Το διακρίνουμε καθαρά αυτό. Θα πρέπει βέβαια να λάβουμε υπόψη μας και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με τη Σερβία δίπλα τους και την ειδική τους κατάσταση που εκεί ισχύει αυτή που τους εμποδίζει να πετύχουν. Ελπίζουμε το αντίθετο όμως να συμβεί στην Ουκρανία, να πετύχουμε εκεί. Να μην χάσουμε βέβαια και την ελπίδα στη Βεσνία Ρεζεγοβίνη. Χρειάζεται να έχουμε αυτήν την άποψη για να μπορέσουμε να πετύχουμε τελικά. Ευχαριστώ. Παρά τις δύσκολες συνθήκες εδώ, κάτω από τις οποίες διεξάγεται η συνάντησή μας, και ότι δεν υπάρχει και πλατιά συμμετοχή, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή κύριο Κλοντή που είναι εδώ για την εισήγησή του. Σίγουρα και στο μέλλον θα σας προσκαλέσουμε και πάλι. Θα διατηρήσουμε μαζί σας τις επαφές και με πολύ πολύ διάθεση θα ακούσουμε και πάλι ειδικότερα σημεία για την Ευλέξ που είναι περίπλοκο θέμα και απαιτείται ακριβώς μια άμεση επέμβαση. Γιατί δυνητικά υπάρχει ένας κίνδυνος. και ε, στο κοσυφοπέδιο και παντού και για την κοινή γνώμη. Η κατάσταση αυτή υπονομεύει τη δική μας αξιοπιστία. Άρα λοιπόν τάχιστα θα πρέπει να αντιδράσουμε σοφά και αποτελεσματικά. Ε, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ναι, μισό λεπτό να δείξω. <laughs> Με συγχωρείτε για το βήχα. μου θυμίζουν ότι η επόμενη συνάντησή μας θα λάβει χώρα τις 20 Νοεμβρίου και βέβαια είστε όλοι καλεσμένοι να παραστείτε. Σας ευχαριστώ. Τέλος της συνεδρίασης.